Καλημέρα σας. Λέω να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε αρκετούς ευρωβουλευτές για να λάβουν το λόγο στο πρώτο σημείο. Καταρχήν να συγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω νεύματα, άρα Ας την εγκρίνουμε. Ανακοινώσει Πρόεδρου υπάρχουν. αυτέ δεν τι γλιτώνουμε. Θα ξαναεπιληφθούμε του διπλού πακέτου και των εκκρεμωτήτων μετά την τριμερή διάλογο τη 14 η Νοεμβρίου. Έκθεση γκοζέ. Έχουμε κάποιε εκκρεμότητε, τρόποι ψηφοφορία στο Συμβούλιο και κάποια τμήματα του, συμβουλ... του Μνημονίου Κατανόηση ό,τι αφορά την πάταξη τη φοροδιαφυγή. Για την έκθεση Φερέιρα Προσπαθούμε να σημειώσουμε πρόοδο στα διάφορα άρθρα και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια σημεία για την τελική πολιτική συζήτηση, όπως ο δικός χάρτης για τα ευρωομόλογα και το Ταμείο Απόσβεσης, το Redemption Fund. Σε ό,τι αφορά την οδηγία κεφαλαϊκών απαιτήσεων και το σχετικό κανονισμό, ε, έγινε εκτεταμένη συζήτηση. Δευτέρα, πρώτη και απόγευμα πήγε μέχρι και το βράδυ για πολλά κρεμή θέματα. Μακροπροληπτική ελαστικότητα για την ρευστότητα των κρατών μελών, προσαρμογέ ε, της ε, αξίας του δανεισμού και υποβλήθηκαν πολλές συντακτικέ τροπολογίες. Θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο αυτή τη βδομάδα εργασίες και ε, θα λάβετε την Παρασκευή την ενημερωμένη συμβιβαστική πρόταση. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει το πρωί της 20 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη το πρωί. Και ας περάσουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, την άγγιση της ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η συγγήτριά μας για το θέμα αυτό είναι η Άννη Ποδήματα, που ήταν και η συγγήτρια για την αρχική έκθεση. Δεν έχουμε δεν πρόκειται για διεκπαιρέωση του έργου, μάλλον για συνέχεια. Έχει το λόγο, Άννη. Ευχαριστώ, Σάρων. Έχει απόλυτο δίκιο ότι εδώ εξετάζουμε τη σύσταση του Κοινοβουλίου προς την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής για μία απόφαση του Συμβουλίου που θα ε, δίνει έγκριση άδεια για την ενισχυμένη συνεργασία σε ό,τι φορά το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο συντρέχουν οι ένομες προϋποθέσεις για την ενισχυμένη συνεργασία, όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Ως προς τη διαδικασία λίγες ε, λεπτομέρειες, μετά τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει έγκριση με ειδική πλειοψηφία για την ενισχυμένη συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει αναθεωρημένη πρόταση επί της ουσίας με βάση την αρχική πρόταση και ελπίζουμε θα λάβει υπόψη και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του περασμένου Μαΐου. Να σας υπενθυμίσω ότι μετά από ένα χρόνο συζητήσεων στις 27 χώρες μέλη με βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε υποβληθεί στις 28 Σεπτεμβρίου του 2011 η Κυπριακή Προεδρία τελικά τον περασμένο Ιούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα συγκεντρωθεί ομοφωνία υπέρ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο μέλλον, οπότε τον Οκτώβριο πριν από ένα μήνα δηλαδή, 11 χώρε μέλη, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εστονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, έστειλαν επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας ε, την θέσπιση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με βάση το κανόνα της ενισχυμένης συνεργασίας. Και όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ από προχθές και η Ολλανδία εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ενισχυμένη αυτή συνεργασία, υπό όρους όμως. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο ήδη έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις, μάλιστα με αρκετά συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα. Ήδη αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ, της προχθεσινής συνεδρίασης. Εκεί έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση για το θέμα αυτό και στα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ αναφέρεται ότι τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε να ληφθεί απόφαση μέχρι το Δεκέμβριο. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη θέσπιση του φόρου από το χρηματοπιστωτικό συναλλαγό στην Ευρώπη και συστηματικά ασκήσαμε πίεση και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Επίσης, στη γνωμοδότησή μας του περασμένου Μαΐου αναγνωρίσαμε τους περιορισμούς που ενέχει μια διαδικασία ομοφωνίας για όλα τα φορολογικά θέματα και μάλιστα επικρίναμε σε πολλές περιπτώσεις αυτούς τους περιορισμούς. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την γνωμοδότησή του τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας για τη θέσπιση ενός φόρου ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εφόσον δεν συγκεντρωθεί ομοφωνία και εφόσον μία ομάδα χωρών επιθυμεί ταχύτερη πρόοδο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν συνεπείς, γι' αυτό και θα ακολουθήσουμε και εμείς ένα συμπλησμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύσταση αυτή, που αφορά, όπως είπα και πάλι, ε, τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, ώστε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, του Δεκεμβρίου να δοθεί έγκριση και να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η συζήτηση της αναθεωρημένης πρότασης επί της ουσίας όμως αυτή τη φορά. Τώρα, για να δούμε τι όροι ισχύουν για την έγκριση της ενισχυμένης συνεργασίας. Με βάση το άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 326 έως 334 ε, περιλαμβάνονται πολλές νομικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέξουν πριν υποβάλει η Επιτροπή την πρόταση για την ενισχυμένη συνεργασία και θα ήθελα να σχολιάσω τις πιο σημαντικές αυτές προϋποθέσεις. Καταρχήν, η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα τομέα που καλύπτεται από τη συνθήκη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 113, που αναθέτει αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εναρμόνιση τη έμεση φορολογία. Άρα πληρείται αυτή η προπόθεση. Επίση, η ενισχυμένη ε, συνεργασία θα πρέπει να είναι ίστατη λύση και όπω είπα, κανένα δεν θα έχει αντίρρηση, ούτε θα αφισβητεί το γεγονός ότι ένα τέτοιο σύστημα στο εγγύς μέλλον δεν πρόκειται να συγκεντρώσει ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών για την επιβολή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επίσης, η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να προωθεί τους στόχους της Ένωσης και να προασπίζει τα συμφέροντά της, ενισχύοντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Και μάλιστα θεωρώ ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πληρεί και αυτέ τι προποθέσει, γιατί θα συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη, ενοποιημένη εσωτερική αγορά, και θα είναι ένα πρώτο βήμα της εναρμόνισης μεταξύ 11 ή και περισσότερων, ελπίζουμε, φορολογικών καθεστώτων. Επί του παρόντος, ισχύουν διάφοροι φόροι επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, διαφορετικοί όμως από αυτόν που προτείνεται τώρα και ισχύουν σε διάφορα κράτη-μέλη και μάλιστα ο ρυθμός τους θα αυξηθεί στο μέλλον, προβλέπετε. Οπότε η εισαγωγή ενός ε, φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε περιορισμένο ρυθμό χωρών με βάση την ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια ουσιαστική ενιαία αγορά. Μια και ο, ένας τέτοιος ενιαίος φόρος θα αποτελέσει το πρώτο επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ αυτών των 11 ή παραπάνω συμμετεχόντων χωρών. Αυτό δηλαδή που θα αποφασίσουν να εισαγάγουν το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτή η κατάσταση αποτελεί, επαναλαμβάνω, το πρώτο βήμα της εναρμόνισης που είναι πολύ ε, καλύτερο από την ισχύουσα κατάσταση που ε, χαρακτηρίζεται από κατακαιρματισμό. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία νομοθετική πρόταση για, τα για το θέμα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πρόκειται για την οδηγία που αφορά τους έμεσους φόρους ε, στο κεφάλαιο και μάλιστα ο FTT συνάδει με το θέμα αυτό, μια και οι πρωτογενεί αγορέ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή. Ε, πέμπτον, η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα πρέπει να υπονομεύει την εσωτερική αγορά, όπω είπα και προηγουμένω. Και επίση, ο φόρος αυτός ε, με βάση την ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να συμβάλλει σε ένα πρώτο επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ των διαφόρων φορολογικών καθεστώτων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μεταξύ των 11 ή και περισσότερων, ελπίζουμε, συμμετεχόντων χωρών, δηλαδή αυτών που θα τον εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι είναι κάπως υποκριτικό να ισχυριζόμαστε ότι ο φόρος επί το χρηματοπιστωτικό συναλλαγών θα υπονομεύσει την εσωτερική αγορά. Γιατί η παρούσα κατάσταση, αυτή η κατακαιρματισμένη, αποσπασματοποιημένη κατάσταση, αποσπασματική κατάσταση είναι αυτή που διακυβεύει και υπονομεύει την εσωτερική αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι το σημείο αφιωτηρίας μας είναι αυτός ο πλήρης κατακαιρματισμός που ισχύει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει καθο... δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε θέσει ως διορία για τις τροπολογίες ε, την 20 Νοεμβρίου, πολύ βραχία προθεσμία. Βέβαια, πρόκειται για αμυγός διαδικαστικό θέμα, πρέπει να δώσουμε τη συνένεσή μας Γι' αυτό και πιστεύω ότι την ενέργειά μας θα πρέπει να την ε, διαφυλάξουμε για τη μεταγενέστερη συζήτηση που θα είναι πολύ σφοδρή επί της ουσίας. Με τη σύσταση πάντως αυτή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ε, την ευθυγράμμιση της ενισχυμένης συνεργασίας με τις συνθήκε και ε, θεωρούμε ότι η ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό είναι ακριβής. Αυτά. Ευχαριστώ, Άννη. Ο Ζαν Πολ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα ομιλώ εκ μέρους της κυρίας Λούλεν λοιπόν, έγινε κοσμήτωρ, πρεσβύτερος του Κοινοβουλίου και θα σας διαβάσω ακριβώς το μήνυμα το οποίο αποστέλει στους συναδέλφους η κυρία Λούλινγκ. Να πω ότι αυτή είναι η θέση της κυρίας Λούλεν Τιμωρούμε λιγάκι εδώ γιατί εγώ την όρισα εισηγήτρια γνωρίζοντας ακριβώς τη μεγάλη αποστροφή που έχει για τον φόρο αυτό και ε, σήμερα καλούμε να διαβάσω αυτό το οποίο θα ήθελε να πει. Πρόεδρε λοιπόν, απούσα ούσα ε, θα ζητήσω από τον συντονιστή μου να μεταφέρει τις απόψεις μου. Οι πολλαπλές συζητήσεις τις οποίες είχαμε γύρω από το φόρο αυτό δεν χρειάζεται φυσικά να επαναληφθούν στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας αδειοδότησης ενισχυμένης συνεργασίας. Ανήκω σε, στους επιφυλακτικούς οι σκεπτικιστές γενικά γύρω από το θέμα αυτό, αν και δεν είμαι κατηγορηματικά αντίθετη. Η πλειοψηφία των βουλευτών λοιπόν εξεφράστη, δεν χρειάζεται να επανέλθω. Να πω όμω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό το οποίο μα ζητείτε στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με την ε, μέγιστη σοβαρότητα γιατί το Κοινοβούλιο παίζει ένα κρίσιμο ρόλο ε, ε, γιατί πρέπει φυσικά να εγκρίνει τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν οι ευρωβουλευτές να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και στον τομέα αυτό που είναι ο τομέας τη φορολογίας. Καλό θα ήταν οι ιδεολογικές διαφορές να αφήσουν τη θέση τους σε συζητήσεις επί της ουσίας που βασίζονται στα γεγονότα και στο δίκαιο. Τρεις παρατηρήσεις, λέγει η κυρία Λούλινγκ. Πρώτη. Η πρώτη αφορά τις επιλογές της διαδικασίας. Η Επιτροπή μας έχει μία πρόταση αδειοδότησης της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα των φόρων για τις χρηματοοικονομικές, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, χωρίς να συνοδεύεται από ένα σχέδιο κειμένου για τον ίδιο το φόρο. Αυτό επί της ε, νομικής ε, πλευράς δεν είναι κάτι το απορριπταίο, αλλά από την άλλη είναι πολύ ενοχλητικό να υπάρχει η αρχή τόσο μακράν ε, από την ουσία. Θα ήθελα να είχαμε ένα προσχέδιο έστω κειμένο. Το να επιτρέψουμε μια ενισχυμένη συνεργασία χωρίς να γνωρίζουμε τις συνέπειες, αυτό είναι κάτι το οποίο με οδηγεί στο να δυσθυμίσω Πρέπει να είστε βέβαιοι συνάδελφοι ότι το Συμβούλιο δεν θα πάρει την απόφαση παρά μόνο όταν έρθει το σχέδιο. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα πιο πριν. Δεύτερη παρατήρηση. Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά μόνο την αρχή. Θα ήθελα όμως επί τη βάση ενός παραδείγματος να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να μας κάνουν να το πιστεύουμε. Η δημιουργία ενός τέτοιου φόρου μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα δύσκολο στη διαχείρισή του ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέχουν και σε αυτούς οι οποίοι ε, είναι αν θέλετε στο περιθώριο, αλλά μέσα στην Ένωση. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αμφισβητήσει την ενία αγορά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εάν η ενισχυμένη συνεργασία η οποία θα δημιουργηθεί οδηγήσει σε μια μαζική μετακίνηση ε, των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε άλλα τμήματα της Ένωσης, αυτό θα είναι δύσκολο να το χωνέψει κανείς. Αν υπάρξουν ε, εξωτοπικές, αν θέλετε, λογικές και ρυθμίσεις, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες οι χώρες οι οποίες δημιουργούν την συνεργασία αυτή επιβάλλουν κάποιες φορολογικές επιβαρύνσεις στα κράτη τα οποία δεν τις επιθυμούν. Συνεπώς λοιπόν το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα τα κράτη εμπλέκονται εδώ και όχι μόνο αυτά τα οποία θέλουν να συμμετέχουν στη συνεργασία. Τρίτη παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να αποφύγει μια σοβαρή μελέτη επιπτώσεων για τις ε, επιπτώσεις ακριβώς, για τις συνέπειες της εισαγωγής αυτού του φόρου σε οικονομικό επίπεδο. Σε δύο μάλλον επίπεδα. Πρώτον, επιπτώσεις στην ενιαία αγορά και δεύτερον επιπτώσεις ανάμεσα στις χώρες οι οποίες είναι μέλη αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας και αυτές που είναι εκτός αλλά επηρεάζονται. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι ε, μέσω αυτής της διαδικασίας ε, θα πρέπει φυσικά να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να θέσουμε ερωτήσεις επί της ουσίας, ερωτήσεις γαλήνιες, για να αποδειχθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα σοβαρό εταίρο ακόμα και στον τομέα της, της ε, Τάδε Εφη Λούλιν. Μπράβο λοιπόν για του φιλελευθέρου. Βολφ. Ο Βολφ δεν είναι εδώ μάλλον. Αντίθετα με τον Ζαν Πολ, ο συνάδελφος μου δεν μου έχει δώσει τίποτα σε έγγραφη μορφή για να σα διαβάσω. Ούτε καν μου μίλησε και μου παρουσίασε τις ιδέες του. Άρα θα σας παρουσιάσω τις δικές μου απόψεις. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ζαν Πολ για την Άστριντ. Αφενός, εξ όσων γνωρίζετε, υποστήριξα την πρόταση υπό τον όρο ότι όλα τα, κράτη-μέλη θα συμμετείχαν. Και όταν κατέστησε σαφέ ότι αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί, τότε είπα ότι θα έπρεπε να τροποποιήσουμε το κείμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πιθανότητα να συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη να ήταν πιο μεγάλη. Και είπα ότι θα έπρεπε για παράδειγμα να κοιτάξουμε τον φόρο για τις μετοχές ε, που επιβάλλονται στην Ηνωμένο Βασίλειο στην παρούσα φάση και να τον τροποποιήσουμε, να τον αυξήσουμε, να τον προσθέσουμε δηλαδή και σε άλλα αξιόγραφα ε, σταδιακά όσο θα αποκτούσαμε εμπειρία. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό ως πρόταση για διάφορους λόγους. Και τώρα βρισκόμαστε στην παρούσα κατάσταση. Κάποιες παρατηρήσεις επιτρέψτε μου. Καταρχάς, θεωρώ ότι Εφόσον το Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την πρόταση αυτή, νομίζω ότι σωστό είναι να υποστηρίξουμε και τα κράτη-μέλη που αποφάσισαν να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα σε πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Ωστόσο, ανακύπτουν μια σειρά από σημαντικά, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Καταρχάς, συμφωνώ με την Άστρετ Ποιο είναι το τελικό κείμενο. Ποιο κείμενο θα εισαγάγουν και θα εφαρμόσουν για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τα κράτη αυτά που επιθυμούν να το εφαρμόσουν. Είναι σημαντικό αυτό. Περιεριζόμαστε στην αρχή του κατοίκου, περιλαμβάνουμε και την αρχή της προέλευσης. Πώς. Τι θα γίνει, ο φόρος αυτός θα εφαρμοστεί και θα ισχύει και για χώρες εκτός των χωρών που τον εφαρμόζουν. Αυτό αφενός. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει μια καλή μελέτη δικτύπου που θα μας καταδείξει με τρόπο πιστικό ποια θα είναι τα, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τις χώρες που θα εφαρμόσουν το φόρο και για τις υπόλοιπες χώρες. Κατά τρίτον, ξέρουμε πού θα καταλήξει τελικά αυτός ο φόρος. Γιατί αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα πιο πολλά κράτη που συμμετέχουν, έχουν ε, διοχετεύσει ε, τα έσοδα στον προπολογισμό τους στην παρούσα Εγώ περίμενα ότι θα διοχετευτεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αν συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι και οι χώρες αυτές θα πρέπει να μεταφέρουν λιγότερα κονδύλια, λιγότερες, ε, λιγότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Και τι γίνεται για τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, για παράδειγμα, από την Business Europe, που, από τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, που ε, δηλώνουν ότι θα μειώσει αυτό το ρυθμό ανάπτυξη ε, στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκφράστηκαν τέτοιε ανησυχίε. Άρα θα έλεγα ότι επί της αρχής, και νομίζω ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι, επί της αρχής λοιπόν συμφωνούμε την προσέγγιση αυτή και υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη που θέλουν να εφαρμόσουν το φόρο αυτό στα πλαίσια ενισχυμένη συνεργασία, τολμηρά και θαραλέα. Δεν λέω, αλλά υπάρχουν ακόμα εκρεμή ζητήματα, στα οποία θα ήθελα μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα για τους πράσινους, η Έμιλη. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την ε, εισηγήτρια. Συμφωνήσαμε για την ε, ταχεία διαδικασία και θεωρώ ότι αυτή η... αυτό το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς και έχουμε μια καλή βάση της 31ης Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται πλέον για μια πρόταση όχι για 27 κρατημέλη, αλλά στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Δεν ε, περιμένω ότι το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει ε, ε, για όλα τα ζητήματα. Να σας πω ότι οι πλευρά περιεχομένου περιλαμβάνονται κάποια στοιχεία στις συντελογικές σκέψεις. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να προσταθούν και άλλα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία από πλευράς μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε τι αποφασίσαμε στις, 31 Μαΐου. Ότι ο φόρος θα πρέπει να ισχύει για όσο πιο πολλά χρηματοοικονομικά μέτρα και μέσα γίνεται. Επίσης, να υπενθυμίσουμε τις τεχνικές βελτιώσεις που έγιναν, προς προσθήκη της αρχής της ασφάλισης και για να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Λούλη, για να αποφύγουμε τη διαφυγή κεφαλαίων, τη φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι αυτό έχει ως σκοπό η αναδιαμόρφωση του κειμένου. Κατά τρίτον, θα πρέπει να αναφέρεται, πιστεύω, ότι θέλουμε να προωθήσουμε ένα καθολικό φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν στα πλαίσια του G20. Τέταρτον, όπως είπε και ο κύριος Κλίνς, Ίσως θα έπρεπε να σχολιάσουμε τον φόρο αυτό ως ίδιο πόρο. Αυτό περιλαμβάνεται στο κουτί το διαπραγματευτικό της Κυπριακής Προεδρίας. Ότι οι χώρες δηλαδή μπορεί να συμβάλλουν με τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να περιορίσουν έτσι τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Και τέλος, Αυτέ είναι κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε να μπουν ε, από πλευρά περιεχομένου στι στις σκέψει. Και βασικά, πολύ σημαντικό είναι να βασιστούμε στην έκθεση της 31ης Μαΐου, η οποία ήταν απόρρια ε, εκτενών συζητήσεων και στην Επιτροπή μας αλλά και σε άλλες επιτροπές. Να πω τώρα δύο λόγια για το Συμβούλιο. Βλέπουμε ότι οι κάτω χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν το φόρο έχουν κάποιες... Ε, ζητούν να περιοριστεί το εύρο εφαρμογή του φόρου. Δεν θα το αποφασίσουμε εμεί αυτό ασφαλώ, αλλά είναι θετικό. Θετική ένδειξη το γεγονό ότι τον εξετάζουν τον φόρο αυτό όλο και πιο πολλέ χώρε. Γιατί θεωρώ ότι όσο πιο πολύ τον εφαρμόζουν, τόσο πιο πολλέ χώρε που δεν τον εφαρμόζουν θα φοβούνται μήπω χάσουν έσοδα. Δηλαδή θα Πρέπει οι Σουηδοί, οι Δανείοι να πληρώνουν φόρους για ένα ευρωπαϊκό, για την ευρωπαϊκή αγορά. Και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές και σε άλλες χώρες. Επίσης άκουσα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον ε, εξετάζει το ενδεχόμενο να αντιταχθεί στο Συμβούλιο. Ευτυχώς δεν χρειάζεται ομοφωνία, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η τάση. Σας καλώ όλους λοιπόν να δείτε τι γίνεται με τις κυβερνήσεις σας και να μην επιτρέψετε να παρεμποδίσουν το σχέδιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουν όσο πιο πολλές χώρες γίνεται. Το καλό είναι ότι στα πλαίσια της ε, ενισχυμένης συνεργασίας μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε χώρα ανα πάσα στιγμή. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι ανοιχτή η πόρτα δηλαδή. Και φυσικά αυτό που θα θέλαμε είναι να συμμετάσχουν όσο πιο πολλές χώρες γίνεται. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το προωθήσουμε αυτό. Για να μην υπάρχουν και περαιτέρω εμπόδια, να μην ε, παρουσιάσει εμπόδια το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω να αναλυθεύουν αυτέ οι φήμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρο. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο από το ECR, από του ε, συντηρητικού, ο Γιούργεν από την ΚΟΕ. Ο Γιούργεν από την ΚΟΕ, ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ο σκιώτη ε, συγητή. Η Μαρίζα ήταν σκιώτη η η Μαρίζα Ματία, η οποία δυστυχώ ασθενεί σήμερα και με παρακάλεσε να μιλήσω εκ μέρους της, αλλά έχει γράψει ένα κείμενο. Αλλά όχι, είμαι, μπορώ να μιλήσω κι εγώ, όπως ο Γιούργεν, να παρουσιάσω και τις ε, δικές μου απόψεις. Ε, υποστηρίζουμε τον φόρο χρηματοοικονομικών αλλαγών και την έκθεση που έχει παρουσιάσει η Ανυποδηματά. Καλωσορίζω λοιπόν και την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι είναι κάτι να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Το συζητάμε εδώ και δύο-τρία χρόνια το θέμα των χρηματοοικονομικών φόρων, των φόρων επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ξέρουμε γιατί, το γιατί είναι τόσο σημαντικό. Στην κοινωνία των πολιτών διακρίνουμε μία σειρά δραστηριοτήτων, αναφορές και άλλες αναφορές από ενώσεις των πολιτών που υποστήριζαν και υποστήριξαν την εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη με αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες που είναι οι εκλογείς μας περιμένουν να συμβεί κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Το προστακούν αυτό. Εγώ από δικής μου πλευράς και αυτή είναι η πλευρά που ε, παρουσιάζει και η Μαρίζα, υποστηρίζουμε την Άννη. Έχουμε όμως κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε. Τα είπε και ο Βούλφ. Να προσέξουμε, να μην καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα πετύχει κάτι διαφορετικό από αυτό που αποσκοπούμε. Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εδώ το θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αυτό το βήμα προκειμένου να δοθεί το μήνυμα προς τους πολίτες ότι δεν περιοριζόμαστε σε συζητήσεις και ότι κάτι πετυχαίνουμε τελικά. Φυσικά και θα επιθυμούσαμε να μην συμμετείχαν μόνο κάποια κράτη-μέλη, να συμμετείχαν όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά είναι γνωστό ότι αυτό πολύ απλά δεν μπορεί να περάσει στην παρούσα φάση. Δεν είναι ρεαλιστικό λοιπόν. Άρα ο μοναδικός τρόπος που έχουμε για να προχωρήσουμε το θέμα αυτό είναι η ενισχυμένη συνεργασία. Το υποστηρίζουμε λοιπόν και ελπίζουμε πραγματικά να μας οδηγήσει παραπέρα αυτό το βήμα. Ε, ευχαριστώ. Τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις ε, και θέλησα να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάπου πίσω βρίσκεται κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω έξι παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε ερωτήσεις που έγιναν. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί επιτάχυνε τις ε, εσωτερικές διαδικασίες λήψη αποφάσεων στέλνοντας ένα σαφές και χειρό μήνυμα ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλουν να γίνουν εμπόδιο στην ενισχυμένη συνεργασία και σε μια ταχεία ε, έγκριση του κειμένου και της θέσπισης του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Χαίρομαι επίσης για το ότι φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, και θεωρεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έγκριση της, του αιτήματος ενισχυμένης συνεργασίας. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μην ξεχνάτε ότι η εναλλακτική λύση ως προς την, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν είναι παντελής έλλειψη φορολογίας αυτής 11 χώρες, αλλά είναι η εφαρμογή 11 διαφορετικών φόρων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αντί για ένα ενιαίο, κάτι που εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέταρτο σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει όντως την πρόθεση να υποβάλει μια πρόταση επί της ουσίας για τον τρόπο εφαρμογής της ενισχυμένης συνεργασίας και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Αλλά τις επιστολές τις λάβαμε μόνο τον Οκτώβριο από τα κράτη-μέλη και μόνο εκεί φάνηκε με σαφήνεια ο στόχος και ε, ο σκοπός, η αποστολή της ενισχυμένης συνεργασίας. Πάντως, σας διαβεβαιώ ότι το σημείο φετηρίας της ενισχυμένης συνεργασίας ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πλησιάζει με την αρχική, στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες προσαρμογές, με κάποιες ε, αλλαγές που κατέσαν απαραίτητες. Πάντως, ε, θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στην έκθεση του ε, Μαΐου, για παράδειγμα, να ενισχύσουμε τα μέτρα για να αποφύγουμε τη μετατόπιση, το θέμα της αρχής της έκδοσης κτλ. Πέμπτο σχόλιο. Για τη μελέτη επιπτώσεων, όπως την ε, χαρακτηρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα, θα υποβάλει μια νέα πρόταση που θα είναι πανομοιότυπη με την αρχική. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε εκ του μηδενό. Ο μηχανισμό θα μείνει σχεδόν απαράλλαχτο και τα αποτελέσματα θα είναι σχεδόν τα ίδια. Αυτό που θα κάνει όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να συμπληρώσει τη μελέτη επιπτώσεων που ήδη έχει καταθέσει, να τη συμπληρώσει με την ανάλυση που έκανε το Μάιο και να προσθέσει μια νέα ανάλυση των επιλογών και των συνεπειών της ενισχυμένης συνεργασίας. Φυσικά αυτά θα υποβληθούν από κοινού με την ε, ουσιαστική πρόταση. Και το τελευταίο μου σχόλιο. Ε, παρόλο που δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδικασίας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η θέσπιση του φόρου από μία μικρή μονομάδα χωρών δεν θα έχει αρνητικές συνέπειε ούτε για τι συμμετέχουσε χώρε ούτε για αυτές που βρίσκονται εκτός της συμφωνίας. Και για να είμαι ειλικρινή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι επιφυλάξει ε, των μη κρατών για το ότι θα του βλάψει αυτή η έλλειψη συμμετοχή. Αν, ε, υποβληθεί, αν θεσπιστεί ένα τέτοιο φόρο ε, σε ορισμένε χώρε, σε καμία περίπτωση δεν θα βλάψει σε, δεν θα βλάψει άλλες χώρες, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη. Ε, ε, και οι διεθνείς εταίροι μας δεν ανησυχούν. Με εκπλήσει λοιπόν που οι μη συμμετέχουσες χώρες θεωρούν ότι θα έρθουν σε δυσμενή θέση σχέση με τις συμμετέχουσες. Σας διαβεβαιώ επίσης ότι ο φόρος αυτός ούτε τις χώρες που θα τον εφαρμόσουν θα βλάψει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει πολύ ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα αποφυγής της μετατόπισης. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο πρότεινε και σχετική τους ενίσχυση. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι με βάση τα αρχικά απορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διαπιστώνεται κανένα οικονομικό πρόβλημα, ούτε κανένα πρόβλημα στην εσωτερική αγορά με την θέσπιση ενός τέτοιου φόρου από περιορισμένο αριθμό χωρών. Όλο Νάρντο. Σύντομα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε μόλις ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Θα συμφωνήσω με την κυρία Ποδηματά στην ανάγκη η οποία υπάρχει να ευνοήσουμε με τον μέγιστο τρόπο την εναρμόνιση τη φορολογική ανάμεσα στις χώρες οι οποίες επέλεξαν την ενισχυμένη αυτή μορφή συνεργασίας. Διαρωτώμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος τον οποίο προοπτικά θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει και αυτό να έχει έναν σημαντικό ρόλο. Τρει ερωτήσεις να θέσω τώρα. Η πρώτη αφορά την ανάγκη, όπως είπα, η οποία υπάρχει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα από τη μία στον φόρο, στην ίσπραξη του φόρου και στον κίνδυνο φόρο αποφυγής από την άλλη. Μήπως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθμίσουμε το ύψος του φόρου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ε, χτυπήσουμε αν θέλετε με αποτελεσματικό τρόπο τις high frequency trading, τις ε, συναλλαγές υψηλής ε, ταχύτητας ουσιαστικά έτσι ώστε να μην υπάρχει φοροαποφυγή και να μην επιβαρύνουμε μόνο τις επενδύσεις και τις συναλλαγές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Τώρα, δεύτερη ερώτηση για αυτά τα οποία είπε ο Βολφ Κλίνγκς. Μου κάνει εντύπωση το ότι μία σειρά κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και η Ιταλική, ενέκριναν ήδη τον εσωτερικό τους νόμο σταθεροποίησης, εξυγίανσης, προβλέποντας και κάποιες ρυθμίσεις για την εισαγωγή του συγκεκριμένου φόρου και πιθανά έσοδα από την εφαρμογή του φόρου αυτού. Νομίζω ότι πρέπει να προηγηθεί μια κάποια εναρμόνιση και μια θα έλεγα κοινά αποδεκτή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη τα οποία θα προχωρήσουν στην επιβολή του συγκεκριμένου φόρου. Τρίτον, για την επιβολή του φόρου στον ε, καθημερινό κύκλο εργασιών ή στις μεμονωμένες συναλλαγές. Αν θα πρέπει να προστίθενται όλα στο τέλος της ημέρας δηλαδή ή θα πρέπει να φορολογείται επιμέρους κάθε ε, συναλλαγή. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της λύσης, της μεμονωμένης συναλλαγής. Και τέλος υπάρχει και άλλο ένα ευαίσθητο αρκετό θέμα, το οποίο αφορά την ε, φορολογική έδρα θα λέγαμε, ενός από τους δύο συμμετέχοντες στη συναλλαγή. Αν θα πρέπει δηλαδή να επιβάλλεται ο φόρος επί τη βάση της φορολογικής διεύθυνσης ή επί τη βάση της εθνικότητας του asset το οποίο γίνεται αντικείμενο συναλλαγής. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να εκφραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν έχω αμφιβολία ότι με τις προσπάθειες που έγιναν από την εισηγήτρια θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα θετικό βήμα. Um, uh, έχουμε 10 λεπτά. Θέλετε να δώσετε κάποιος, κάποιο σχόλιο σε αυτά τα οποία είπε ο προηγούμενος ομιλητής, αλλιώς θα δώσω το λόγο στην Άννη. Ναι, έχουμε σχεδιάσει την πρόταση έτσι ώστε η υψηλή ταχύτητα συναλλαγές να καλύπτονται. σχετικά τώρα με τις δαπάνες. Ίσως να έχει υπάρξει μια παρανόηση του τι ε, εννοεί ιδίους πόρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λέμε ότι το τμήμα του FTT πρέπει να πηγαίνει μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αυτό όμως σημαίνει ότι στο τέλος Όταν γίνει δεκτή η πρόταση ε, ε, για τους ιδίους πόρους, ε, τα χρήματα που θα έχουν συλλέξει τα κράτη-μέλη από το φόρο αυτό θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Δεν πρόκειται. Περνάνε μεν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά δεν οδηγούν στην αύξηση του προϋπολογισμού. Εφόσον μπορούν ε, να συμφωνήσουν οι 11 χώρες, ε, τότε ήδη από το 2014 μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και μπορούν για το 2014 να το λάβουν υπόψη στις προβλέψεις τους για τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει για το 2013 όμως. Τώρα για τον κατάλογο των κριτηρίων. Όταν δεν εκπληρούνται το πρώτο κριτήριο, τότε θα εξετάζεται το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κτλ. Εμείς έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ε, μια συγκεκριμένη σειρά. Τώρα, αν οι χώρες θέλουν να ταξινομήσουν με διαφορετικό τρόπο τα κριτήρια αυτά, Αυτό ε, είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ είναι στόχος της ενισχυμένης συνεργασίας και θα καθορίσει τα πόσα χρήματα θα δίδονται, εν πάση περιπτώσει και σε ποιες χώρες. Άννη, έχει το λόγο. Thank you, Sharon. Ευχαριστώ, Σάρον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις τους παρόλο που μερικές θεωρώ ότι δεν ε, έχουν θέση στη συγκεκριμένη σύσταση, γιατί η σύσταση αυτή επικεντρώνεται μόνο στην ε, ε, έγκριση των κανόνων, στην αδειοδότηση των κανόνων της ενισχυμένης συνεργασίας, δεν αφορά την ουσία. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να αποσυνδέσουμε τη συζήτηση επί της διαδικασίας από τη συζήτηση επί της ουσίας. Έχω δύο σχόλια, Σάρων θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια που μας διάβασε ο Ζαμπόλ Κοζές ε, εκ μέρου της κυρίας Λούλινγκ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την ε, αποσύνδεση της διαδικασίας έγκρισης ε, της ενισχυμένης συνεργασίας από την ουσία της ενισχυμένης συνεργασίας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που έπρεπε να δώσουμε την ε, συνένεση μας, την κατάθεσή μας για την ε, έγκριση μιας ενισχυμένης συνεργασίας, έτσι κάναμε. Δηλαδή πρώτα ασχολούμαστε με τη διαδικασία και αξιολογούμε κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι νομικές προϋποθέσεις της α, ε, ενισχυμένης συνεργασίας και μετά επισερχόμαστε στην ουσία. Άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, ανέκαθεν αυτή τη διαδικασία εφαρμόζαμε. Ε, ευχαριστώ την Έμιλη ε, για τις προτάσεις που έκανε για τους κατοίκους και εγώ αυτό επιθυμώ, ε, να δημιουργηθεί μια συνένεση και να ενισχυθεί αυτή η θέση. Έχω αμφιβολίες ε, για το θέμα των ιδίων πόρων όμως. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δημιούργησε πολλές δυσκολίες και στις προηγούμενες μας συζητήσεις. Επί της γνωμοδοτήσεως δηλαδή που είχαμε δώσει τον περασμένο Μάιο για την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι εξακολουθεί να υπάρχει διάσταση απόψεων για το θέμα των ιδιών πόρων, οπότε θα είναι αρκετά επίμαχο το θέμα. Πάντως, υπενθυμίζουμε την ανάγκη για έναν ευρύ φόρο επί το χρηματοπιστωτικό συναλλαγών, την ανάγκη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη θέσπιση ενός ε, γενικού φόρου, παγκοσμίως δηλαδή, ενός ε, παγκόσμιας εφαρμογής φόρου ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προθυμία της να εστερνιστεί τις τι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βελτιώσει την αρχική της πρόταση. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι θετικά. Τέλος, το θέμα της μετατόπισης και οι ανησυχίε ω προς την εξοδαφικότητα και την μετατόπιση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν μερικοί που ήταν ανέκαθεν επιφυλακτικοί απέναντι στην εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και θεωρώ ότι χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα της ε, ανησυχίας ε, για, ε, για τη μετατόπιση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τώρα φαίνεται ότι μετακινούνται προς ένα άλλο πρόβλημα και την ανησυχία τους για την εξοδαφικότητα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικό και δεν είναι και πολύ λογικό. Όσοι φοβόνταν ότι η εισαγωγή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα οδηγούσε σε μετατόπιση, σε μετεγκατάσταση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα βλέπω ότι φοβούνται ότι η ενισχυμένη συνεργασία για τον χρηματοπιστωτικό φόρο θα είναι τόσο επιτυχημένη που με την εξοδαφικότητα ε, θα οδηγήσει σε μετατόπιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θεωρούν δηλαδή ότι ο φόρος αυτός θα είναι τόσο επιτυχημένος και τόσο στεγανός που θα ε, δημιουργήσει σημαντικό κέρδος και θα αποφύγει την, τον κίνδυνο της μετατόπισης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και προσβλέπουμε με αδειμονία στην αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην μελέτη των επιπτώσεων. Ε, θεωρώ ότι θα τα καλύψει όλα αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη πρόταση και προς το παρόν το συμπέρασμα που μπορώ να συνάγω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να τηρήσει τη θέση και να μείνει στη θέση που έχει λάβει μέχρι τώρα για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να δώσει τη συγκατάθεσή του για την έγκριση της ενισχυμένης συνεργασίας. Αυτά και ευχαριστώ Σάρων. Σε ευχαριστούμε Άννη. Έχω κάποιες ανακοινώσεις τώρα επί της διαδικασίας. Στις 26 Οκτωβρίου οι συντονιστές της ΕΚΟΝ αποφάσισαν να εφαρμόσουμε ένα fast track χρονοδιάγραμμα στη διαδικασία συγκατάθεσης για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου του 2012. Επίσης, οι συντονιστές απέφθαιναν έκκληση ώστε ε, να φροντίσουν οι συντονιστές και οι ηγετές και συγγήτρια ώστε να μην καταταθούν πολλές τροπολογίες και ε, να εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, μόνο στα αγγλικά, να αποφύγουμε τις μεταφράσεις για να προλάβουμε το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, οι τροπολογίες θα πρέπει να αφορούν μόνο τις τιολογικές σκέψεις ή μόνο την παράγραφο 1, ε, προκειμένου να γίνει αρνητική συγκατάθεση. Μόνο συγκατάθεση ή απόρριψη μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την πρόταση. Επαναλαμβάνω, ε, επίσης, ε, τροποποιήσεις για τις θεωρώντας μόνο μπορούν να γίνουν και για δεν μπορούν να γίνουν ε, παρά μόνο γραπτός με χειρόγραφα με τον παραδοσιακό τρόπο. Η προθεσμία λίγη στις 5 το απόγευμα στις 20 Νοεμβρίου και παρακαλώ μόνο στα αγγλικά επιτρέπετε να καταθέσετε τροπολογίες. Την επόμενη Τρίτη, δηλαδή 20 ε, Νοεμβρίου μέχρι τις 5 το απόγευμα, μόνο στα αγγλικά. Θα τις εξετάσουμε στις 28 Νοεμβρίου, θα ψηφίσουμε στις 29 Νοεμβρίου και όπως είπα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αυτή τη σύσταση σας ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ και την Άννη. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τον Τόμας Βίζερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για την ε, Στατιστική Διακυβέρνηση. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με βάση την τέταρτη ετήσια έκθεση της ΕΣΓΑΠ, του Συμβουλευτικού Αυτού Φορέα δηλαδή, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, τα στατιστικά στοιχεία έχουν αρκετή σημασία για την Ευρωζώνη Ελπίζω λοιπόν να παραμείνουν οι συνάδελφοι γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και αν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν παρακαλώ χωρίς φασαρία. Okay. Um, so thank you very much. We, we now have an hour uh, in which to discuss statistics. Έχουμε λοιπόν μία ώρα στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε τέτοια θέματα στατιστικής. Θα δώσω το λόγο στον Τόμας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε αυστηροί σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Δηλαδή μπορεί το κοινό να μας ακούσει και να μας δει. Ο Τόμας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εννοείται ότι έχουμε μέχρι μία ώρα στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο συνεκτικός γίνεται. Είμαι εδώ να σας μιλήσω λοιπόν για την τέταρτη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για την διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής, που ε, ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια για να παρουσιάσει ανεξάρτητη επισκόπηση σε ό,τι αφορά το στατιστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ε, υποδείξατε ήδη πρόεδρε αυτό έχει τις ρίζες του κάπου στην Ευρωζώνη αλλά πέρα από αυτό θεωρώ ότι η επισκόπηση για θέματα στατιστικής και του πώς προκύπτουν τα στατιστικά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε έχετε διαβάσει είτε όχι την έκθεσή μας, δεν ε, θα συγχυστώ άμα δεν την έχετε διαβάσει. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω διαβάσει διαφόρες εκθέσεις και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας και έχω την αίσθηση ότι σκοπός μας είναι αμφότεροι να παράγουμε εκθέσεις που θα βοηθούσαν να βρεθούν ευρωπαϊκές ε, λύσεις. για να έχουμε καλύτερη θεώρηση των ζητημάτων αυτών. Στις ε, καθημερινές μου εργασίες ασχολούμαι με θέματα οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης των 27, αλλά κυρίως με απασχολούν και οι οικονομικές πολιτικές των 17 κρατών μελών που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Να σας διαβεβαιώσω ότι πολλά ζητήματα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι σήμερα ξεκινούν από το πώς καταρτίζονται τα στατιστικά στοιχεία, πώς οργανώνονται οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, πώς σχετίζονται με την πολιτική και τις κυβερνήσεις και πιστεύω ότι το σύστημα πλέον έχει καταστεί πιο διάφανες και πιο αποτελεσματικό. Δεν έχουμε ωστόσο πετύχει όλα όσα θα θέλαμε να έχουμε πετύχει και θα έπρεπε να έχουμε πετύχει. Να κοιτάξω λοιπόν τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ουδέτερα μέσα, τα οποία όμως θα πρέπει να αποτελούν τη βάση και τα αποτελεστικά στοιχεία μιας καλής πολιτικής και όχι αντίστροφα. Όχι να αποφασίζουμε πρώτα ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική και μετά να προσπαθήσουμε να την υποστηρίξουμε με στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι θεωρητική μόνο αυτή η παρατηρήση. Το έχω δει να συμβαίνει και στην πράξη τα περασμένα έτη. Προκειμένου λοιπόν να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι, τους οποίους καλείται να εξετάσει ο συμβουλευτικός μας φορέας. Αφενός λοιπόν, καταρχάς αντιμετωπίζουμε ζητήματα διακυβέρνησης. Να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία. Η επαγγελματική ανεξαρτησία. Μία αρχή που ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αρθών Πρακτικών. Έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία εξετάζουμε, όπως για παράδειγμα ο συντονιστικός ρόλος των, ευρωπαϊκών, των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αυτό είναι δεδομένο στις καθημερινές πρακτικές, αλλά δεν είναι απόλυτα. Εξετάζουμε ζητήματα επισκόπησης. Ζητήματα που αφορούν το ρόλο διορισμού ανώτατων στατιστικών σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάμε πώς ε, λειτουργούν αυτοί που παράγουν τα στατιστικά δεδομένα και οι οντότητες με τις οποίες συνδέονται. Παραδοσιακά τα Υπουργεία διαδραματίζουν το ρόλο αυτό και συγκεκριμένα τα Υπουργεία Οικονομικών. Θέματα ίσης πρόσβασης στα στατιστικά δεδομένα επίσης. Ένα δεύτερο ζήτημα που μας απασχολεί και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε πολλές περικοπές στις οικονομικές δαπάνες είναι η σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας και τους πόρους. Κατά πόσο δηλαδή δαπανώνται αποδοτικά και αποτελεσματικά οι πόροι. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των στατιστικών υπηρεσιών είναι καθοδικά, καθοδική και σε ονομαστικούς όρους σε κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης στους τομείς αυτούς, αλλά ως τώρα η εξοικονόμηση αυτή δεν έχει γίνει μέσω μεταρρύθμισης, αλλά μέσω περικοπών. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου μπορεί να γίνουν περικοπές και αυτό θα το θίξω και αργότερα. Τέλος. εξετάζουμε τα μελλοντικά μας σχέδια, τα μελλοντικά σχέδια σε ό,τι αφορά το επόμενο έτος και σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τον κώδικα ορθοπρακτικών. Για να σας παρουσιάσω κάποια από τα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικά. Ένα από αυτά είναι η επαγγελματική ανεξαρτησία. Η επαγγελματική ανεξαρτησία έχει να κάνει με διάφορες πτυχές. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των εθνικών στατιστικών ε, οργανώσεων, το πώς σχετίζονται με την πολιτική και με τα αρμόδια υπουργεία. Ο δεύτερος τομέας, η δεύτερη πτυχή, έχει να κάνει με, με τον διορισμό και την καθαίρεση των επικεφαλής των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Θα πίστευε κανείς ότι το έτος 2012 αυτό δεν αποτελεί ζήτημα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καθαίρεση των επικεφαλής εθνικών στατιστικών υπηρεσιών έχει συμπέσει με εθνικές εκλογές. Φυσικά είμαστε σίγουροι ότι αυτό ήταν απόλυτα συμπτωματικό και δεν είχε να κάνει τίποτα με τις εκλογές και με το εκλογικό αποτέλεσμα πόσο μάλλον, αλλά θεωρώ ότι η ανεξαρτησία στην επιλογή των επικεφαλής στατιστικών υπηρεσιών είναι εγγυημένη θεωρητικά. Αλλά πιστεύω ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν λόγοι που μας οδηγούν να υποθέσουμε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα οδηγούν στο να αντικατασταθεί ο επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μπορεί η διάδοχοι να είναι πάρα πολύ ικανή. Αλλά προφανώς δημιουργούνται ερωτηματικά και σε ό,τι αφορά την πολιτική συμμόρφωση με θέματα στατιστικής. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι η παραγωγή στατιστικών στοιχείων και η επιλογή της ανάλογης μεθολογίας των ε, πηγών ε, στατιστικών και της διανομής θα πρέπει να μην υπόκεινται σε πολιτικές επιρροές. Αλλιώ κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων κάποιες βραχυπρόθεσμες πολιτικές θα αποκρύψουν ουσιαστικά κάποιες εξελίξεις πολιτικές καθόλου ευνοϊκές. είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να ελέγχουμε. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να εκλεπτύνουμε κάπως, ιδιαίτερα στα κράτη τα οποία είναι με ομοσπονδιακό τρόπο δομημένα είναι η λειτουργία και ο συντονισμός ε, των ε, στατιστικών αρχών. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ενισχυθεί και με νομοθετικές αλλαγές γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο οι οποίες όμως ε, να ακυρώνονται από κάποιες άλλες κεντρόφυγες σε ομοσπονδιακό. για να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της εποπτείας θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα συμβούλια σε εθνικό επίπεδο για την σωστή εφαρμογή του κώδικα πρακτικούς που θα έχουμε προτείνει που θα πρέπει να αποτελούνται όχι μόνο από εκπροσώπους της ίδιας χώρας, αλλά και από συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, από την Eurostat, που θα μπορεί να εκπροσωπούνται στα συμβούλια αυτά. Αυτό θα έχει και βραχυπρόθεσμες ποιοτικές ε, επιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε ένα δρόμο ανάπτυξης με τελικό στόχο τις καλύτερες στατιστικές. Το θέμα της ανεξαρτησίας των προσλήψεων απολύσεων, ίσως μόνο προσλήψεων αυτών των αρχών και των μελών αυτών των αρχών. Αν έχουμε υπερβολικούς αριθμούς κανόνων θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει κανείς την αποχώρηση ενός διαχειριστή, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μέτρα πιο σύντομα και μιας και δεν είναι και κάτι τόσο σημαντικό. οι σχέσεις ανάμεσα στις στατιστικές αρχές και τις υπεύθυνες διοικητικές αρχές επίσης είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί. Αυτές είναι οι συστάσεις τις οποίες κάνουμε. Τώρα για, τις, ε, για τους πόρους και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχει τάση να βλέπει ο καθένας τον εαυτό του με διαφορετικό τρόπο και να λέει ότι στο δικό μου τομέα αρμοδιότητας δεν μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, τη μεγαλύτερη δυνατή αυτό που κάνω. Κανένα κράτο μέλος, κράτος μέλος συγγνώμη, μέχρι τώρα δεν μου έχει πει ότι ένα διοικητικό του κομμάτι πράγματι παραδέχεται ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και κατανοούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια κάποια μείωση. Από την άλλη οι στατιστικοί δέχονται ότι όσο μειώνονται οι προϋπολογισμοί στα κράτη-μέλη, οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να ανταποκατοπτρίζουν και μία μείωση στην παραγωγή στατιστικών. Βλέπουμε ποιες είναι οι χώρες στις οποίες ε, οι περικοπές αυτές είναι άνω το μέσου όρου. Βλέπουμε σε κάποιες από τις λεγόμενες νέες χώρες. Αλλά οι μειώσεις αυτές είναι μικρότερες σε κάποιες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εσωτερικό της ζώνης ευρώ θα έλεγε κανείς ότι σε επίπεδο συγκεκριμένων αριθμών κάποιες φορές οι αμοιβέ διαπιστώνεται ότι έχουν αρχίσει να μειώνονται και μερικές φορές η τακτική είναι να μην αντικαθίστανται οι, οι υπάλληλοι οι οποίοι αποχωρούν ή συνταξιοδοτούνται. Στον τομέα των στατιστικών υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κανείς πιο αποτελεσματικό στη χρήση των στατιστικών, να χρησιμοποιήσουμε την κρίση δηλαδή έτσι ώστε ε, να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία να μην υπάρχει επικάλυψη της χρήσης των στατιστικών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, να υπάρχει σωστή ανταλλαγή μικροδεδομένων, να διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες, Εγώ έχω σαν παράδειγμα ασχοληθεί με το θέμα της διπλής χρήσης στατιστικών δεδομένων από διοικητικές υπηρεσίες στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών εμπορικές στατιστικές. Δεν έχουμε κάνει ακόμα βήματα προόδου σημαντικά και αυτό οφείλεται ουσιαστικά σε μία σκλήρινση θα έλεγα των διοικητικών υπηρεσιών όπου μερικές φορές τα πολιτικά συμφέροντα είναι αυτά τα οποία επιτέλους ορίζουν. Μερικές φορές η ανταλλαγή μικροδεδομένων και η χρήση διοικητικών δεδομένων σε ορισμένες χώρες ε, γίνεται με πολύ περιορισμένο τρόπο λόγω του θέματος της προστασίας των δεδομένων αυτών. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου η βασική αρχή, αρχή της εμπιστευτικότητας φυσικά και του απορρίτου γίνεται ιδιαίτερο σεβαστή. Δεν είμαι βέβαιος ότι όμως αυτές οι σκέψεις, αυτές οι εκτιμήσεις ε, είναι τόσο χρήσιμες έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας. Έχω την αίσθηση ότι αν δούμε το θέμα με πιο αποτελεσματικό, προληπτικό βέβαια τρόπο, θα καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, το οποίο θα μειώσει και την ανάγκη πόρων που αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη μας, οι χώρες μας σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε επίπεδο Eurostat υπάρχουν ε, προβλήματα πόρων, ε, ε, εσόδων και αυτό δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά και κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πάντως υπάρχουν λύσεις μέσω καλύτερης συνεργασίας, μέσω σωστότερης χρήσης των δεδομένων, να γίνουμε ένα μεικτό, ένα κοινό στατιστικό σύστημα των 27 χωρών και όχι απλά ένα συγκερασμός απλώς των διαφορετικών στατιστικών αρχών με τη Eurostat. Η Eurostat κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη και πιο αποτελεσματική και ευρωπαϊκή. Ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και θα τελειώσω είναι τα θέματα της εμπιστοσύνης αν θέλετε και πώς αυτά βγαίνουν προς τα έξω, πώς τα μέτρα των πολιτικών και των στατιστικών έχουν ένα κοινό στόχο να υπάρχουν αξιόπιστες και έμπιστες στατιστικές. Η Eurostat έχει υπογράψει μια τέτοια δήλωση και η Ελλάδα επίσης είναι μια απαραίτητη αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στο στόχο παραγωγής αξιόπιστων στατιστικών και αυξάνοντας ε, την συνειδητοποίηση ε, του κόσμου για τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι στατιστικές αυτές. Και δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται περισσότερο να δουν πώς γίνεται η παραγωγή να το κάνουν. Βέβαια, οι 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κάνει κανένα αποφασιστικό βήμα για την υπογραφή αυτής της ανάληψης υποχρέωσης για την αξιοπιστία των στατιστικών τους, παρότι είναι συμπεφωνημένος ευρωπαϊκός στόχος. κάθε επιρροή την οποία μπορεί να έχετε και από την εμπειρία μου ξέρω ότι έχετε τεράστια επιρροή στον τομέα αυτό, της δήλωσης δηλαδή για την αξιοπιστία, θα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Γιατί αλλιώς ναι, μεν πιστεύουμε ότι η πολιτική πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, τα στοιχεία όμως αυτά πρέπει να είναι αξιόπιστα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι αξιόπιστα, πρέπει να βελτιωθούν και αυτοί που τα παράγουν, που τα συνθέτουν θα πρέπει να είναι ελεύθεροι κάποιων βραχυπρόθεσμων πιέσεων και περιορισμών. Μακρηγόρησα, είπατε όμως ότι είχαμε σχεδόν μια ώρα στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Δεν είχαμε και πάρα πολλά μέλη. Εγώ φα... φανταζόμουν ότι θα ήσασταν ικανός ακόμη και τα στατιστικά στοιχεία να μας τα παρουσιάσετε με συναρπαστικό τρόπο. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις, αλλιώς να θέσω τις δικές μου πρώτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα των αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, όχι μόνο στην τελευταία, αλλά και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και εγώ και ο αντιπρόεδρος ε, Τσικλούνα ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Είχαμε όμως αναθεώρηση του κανονισμού 223 του 2009 και μάλιστα ε, την Παρασκευή λίγη και η σχετική θεωρία για την κατάθεση των τροπολογιών. Οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε αυτό με το τελευταίο σας σχόλιο ή θέλετε κάπου να ασκήσουμε επαφή, ε, ε, πίεση σε σχέση με άλλα σημεία της έκθεσης, γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Τώρα, σε σχεση με αλλα με τις έκθεσεις, γιατι και εμας μας ενδιαφερει να βελτιωθει η ποιοτητα των στατιστικων στοιχειων τωρα σε σχεση με τον κανονισμό αυτό, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ε, ανάμειξη της, του ΕΣΓΑΠ στη διορισμό του διευθυντού της Eurostat. Φαντάζομαι κάποια ανάμειξη είχατε σε αυτή τη διαδικασία επιλογής ή όχι. Με ενδιαφέρει το κατά πόσο και ο δικός συμβουλευτικός φορέας στην, στο διορισμό του διευθυντού της Eurostat. Στο εξαπλό πακέτο είχαμε συμπερίληψη του σημείου αυτού. Βέβαια είχαμε στο έλεος μας στα κράτη-μέλη και ήταν εσκεμμένο αυτό το, αυτή η κίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια υπάρχει πολιτικός σύνδεσμος με το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Και επίσης μιλήσατε για την ανάγκη ανεξάρτητων στατιστικών υπηρεσιών και μεγαλύτερη διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των ομοτήμων. Και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα, μιλήσατε για τις εισαγωγές-εξαγωγές. Και είναι ενοχλητικό όταν συγκρίνουμε α, το ότι πιστεύουν ότι εισάγουν και εξάγουν οι χώρες μέλη και αν το συνδυάσουμε, αν διασταυρώσουμε τα στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι αυτά που πιστεύουν ότι εξήγαν και εισήγαν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. μερικές φορές δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη την πορεία του προϊόντος ε, και δεν ταιριάζουν τελικά τα στοιχεία όταν προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε. Και δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια διακριτική ευχαίρεια μεταξύ των κρατών και τέτοιες διαφορές για το τι συνυπολογίζεται στο ΑΕΠ. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά το ίσα 2010, θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και να δούμε τελικά τι θα γίνει με το ισοζύγιο των πληρωμών. Άλλωστε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Η μεθοδολογία της Eurostat λαμβάνει υπόψη και τις ενδεχόμενε υποχρεώσεις και είναι αρκετά διαφανής αυτή η διαδικασία. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Και η Σοφή Ιντβελτ μπορεί να θέσει ερωτήσεις. Βλέπω να κάνει νεύματα, οπότε φαντάζομαι κάτι θέλει να ρωτήσει. Δύο σύντομες ερωτήσεις, γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένοι με το θέμα. Μόλι από πέρυσι άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό, γιατί ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν βαρετά τα στατιστικά στοιχεία. Ε, και από τη στιγμή που έπαψε να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο, προσπάθησα να ε, το ξεχάσω όσο γινόταν. Αλλά βλέπω ότι αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία τα στατιστικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό που κάθε φορά που έχουμε συζήτηση για τα θέματα αυτά έχω την αίσθηση ότι προστίθενται νέοι κανόνες, νέες συμφωνίες, νέες διατάξεις, αλλά το μήνυμα είναι το ίδιο, ότι η εφαρμογή είναι ελλειπής, ανεπαρκής. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί έχουμε πληθώρα αποφάσεων και όχι καλή εφαρμογή. Πριν από ένα χρόνο ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την αξιοπιστία των ισπανικών στατιστικών στοιχείων τι έγινε, διαλευκάνθηκε αυτό το θέμα, είναι πια αξιόπιστα τα ισπανικά στατιστικά στοιχεία. Γιατί βλέπω να μην μας απασχολεί πια αυτό το θέμα. Και δεύτερη ερώτηση, πιο συγκεκριμένη, αναφερθήκατε και στο θέμα των κυρώσεων στην έκθεσή σας. Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που κράτη-μέλη εμφανώς χειραγώγησαν ή εσκεμμένα ε, δημοσίευσαν ανακριβή στατιστικά στοιχεία. Και αυτή είναι μια ιδέα και του εξαπλού πακέτου. Να επανέλθουμε στην παλιά προσέγγιση, όπου τα κράτη-μέλη μεταξύ τους επιβάλλουν κυρώσεις. Εμείς θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για επιβολή των κυρώσεων. και μόνο με δική πλειοψηφία να, να, να μπορεί το Συμβούλιο να τρέψει μια τέτοια πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν χρήζεται τη προσοχή. Δεν α, συγκεντρώνει μάλλον τη δεωσα προσοχή. Μάλιστα, κάτι άλλο. Τόμα. thanks very uh, Να ξεκινήσουμε με κάποια ζητήματα τα οποία είναι τα πιο σχετικά, αν θέλετε, με τη δική μας ε, εργασία και με το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό 23. Από την έκθεσή μας, αυτό που θεωρώ ότι ακολουθεί το σχέδιο έκθεσης που διάβασα, είναι το εξής. Η έκκληση να συνυπογραφούν οι δεσμεύσει ε, περί αξιοπιστίας από τα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, μία πρόταση να κινηθούμε προς ανεξάρτητα συμβουλευτικά σώματα που θα αποτελούνται και θα εκπροσωπούν ευρωπαϊκά και όχι εθνικά συμφέροντα. Θέματα διορισμού των επικεφαλής των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, έχω δει ότι περιλαμβάνονται αυτά στην έκθεση. Θα πρέπει να καταστούν ωστόσο λειτουργικά όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί κάθε κρατός μέλος με το οποίο ενδεχομένως να έρθει σε επαφή θα σας πει ότι ασφαλώς και είναι ανεξάρτητα τα σώματα αυτά. Προς... Προφανώς. <coughs> Mm, Yeah, yeah. I'll be on the warpath again. Yeah, I just get going, get going. <laughs> um, so I think that. Αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να τα κοιτάξουμε ως προτάσεις άμεσες. Ειλικρινά, να σας πω, μου προκάλεσε έκπληξη σχετικά, ο, ο ρόλος που κλήθηκε να διαδραματίσει ο συμβουλευτικός μας φορέας σε ό,τι αφορά τον επικεφαλής της ε, Eurostat. Και θεωρώ ότι αυτό απέχει παρασάγκα από, από την εντολή μας και από αυτό που θα έπρεπε να περιέχει η εντολή μας. Σε ό,τι αφορά το ελληνική στατιστική υπηρεσία και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της, όχι μόνο το Γιούρα αλλά και de facto από κάποιες πολιτικές επιρροές. υπάρχουν διάφορες υποδειγματικές διατάξεις σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την διορισμό των ε, συμβουλίων στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις περί αξιοπιστίας, διαπιστώνω ότι υπάρχουν ανησυχίες από κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά και πρακτικές που είναι παρόμοιε με αυτέ τη Ελλάδα. Κάποια άλλα ζητήματα που δεν σχετίζονται τα πιο πολλά εξ αυτών άμεσα με την εντολή του συμβουλευτικού μας φορέας. Νομίζω και πρέπει να σας πω ότι η ενασχόληση με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις τις απρόπτες contingent liabilities αποτέλεσε θέμα που με απασχόλησε τακτικά στα πλαίσια και τη συνθήκη του Μάστρεχτ, όπου έγινε η μετάβαση από τις υποχρεώσεις στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Ε, Το θέμα λοιπόν είναι ποιος είναι ο κίνδυνος, ο εκτιμόμενος κίνδυνος για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Αυτό είναι υποκειμενικό στοιχείο. Άρα, ποτέ δεν θα είναι εξίσου αξιόπιστα τα στοιχεία για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις όπως ε, τα στοιχεία για το χρέος για παράδειγμα. Δεν είναι εξίσου αντικειμενικά, αλλά σημειώνουμε καλή πρόοδο, ίσως όχι τόση όσο θα έπρεπε, αλλά σημειώνεται πρόοδο. και όλο και πιο σημαντικό γίνεται καταρχάς να οριστούν οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, κατά δεύτερον να βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η κατάρτιση πολιτικής είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρα, γιατί η κατάρτιση πολιτικών ε, για την οικονομία, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, έχει γίνει αυτοματοποιημένη, αν θέλετε, και δεν ακολουθεί τόσο πολύ ε, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις στην διακριτική ευχέρεια, των κρατών μελών. Και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά σίγουροι ότι ακολουθείται μια διαδικασία που θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές χρηματοοικονομικές πολιτικές, θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας ανεξάρτητης με καλό προσωπικό, με καλές διασυνδέσεις και ότι η διανομή των στατιστικών τομέων αυτών δεν οθεύτηκε από, άλλες, ε, από άλλα στοιχεία. Να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να δώσω παραδείγματα από πάρα πολλά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ε, η εισαγωγή στον τρίτο στάδιο επίπεδο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απασχολούσε και η ανακατάταξη απασχολούσε πιο πολύ τους πολιτικούς παρά τους οικονομολόγους. Το θέμα των καλών στοιχείων, όπως είπατε και εσείς, των αξιόπιστων στοιχείων, δεν περιορίζεται μόνο σε εθνικό επίπεδο και αναφερθήκατε στη, στα ισπανικά στατιστικά δεδομένα. Η Eurostat, βέβαια θα πρέπει να μιλάω εκ μέρους της Eurostat, ξεκίνησε μια σειρά επισκέψεων και διαβουλεύσεων, όχι μόνο με εθνικές αρχές, και θα πρέπει να γίνει μια εξακρίβωση των στοιχείων ε, του ελλείμματος, ε, του χρέους και άλλων ε, συνιστοσών σε περιφερειακό και μερικές φορές ακόμη και σε δημοτικό τοπικό επίπεδο. Και στην περίπτωση της Ισπανίας τα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο ήταν γενικώ αξιόπιστα. Κάποιες αποκλήσεις που σημειώθηκαν από θέματα, για θέματα προσαρμογής ε, δημοσιονομικής δεν ήταν τόσο τεράστιες ε, σε εθνικό επίπεδο. Αλλά το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αφενό και τα συστήματα ε, κοινωνικών ασφαλίσεων αφετέρου μας προβληματίζουν σε πολλά κράτη-μέλη και σε μερικά εθνικά συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων αρχίζουν και συσσωρεύονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ε, κάτι που δεν ε, βαρύνει μόνο τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά δείχνει παρόλα αυτά ε, τις πιέσεις που υπάρχουν στο σύστημα, κάτι που μπορεί μελλοντικά να αποδειχθεί ακόμη πιο προβληματικό. Θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω ότι η ανταλλαγή μακροδεδομένων μεταξύ των εθνικών στατιστικών Ινστιτούτων είναι το θέμα που παρουσιάζεται μεγαλύτερα κενά ε, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ε, παραγωγής πιο αξιόπιστων και ακριβών στοιχείων. Εκεί είναι που χωλένουν τα πράγματα. Οπότε και ελπίζω ότι ότι με το καλό σε ένα χρόνο θα ξανάρθω για να σας παρουσιάσω την πέμπτη της έκθεση του συμβουλευτικού μας Φορέ. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε σημειώσει ε, πρόοδο σε πολλά θέματα και ε, αυτές οι προσπάθειες και οι πρόοδοι αν έχουν γίνει θα οφείλονται όχι μόνο στα στατιστικά, στις στατιστικές φορείς αλλά και χάρη στις δικές σας ε, συμβουλές, προσπάθειες και συνεισφορά. Ο Τόμας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα στον κύριο Βίζερ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε συχνά ότι θέλουμε πιο πολύ Ευρώπη, όχι μόνο Ευρώπη υπό την έννοια της κεντρικής διοίκησης, όχι θέλουμε να λαμβάνονται πιο πολλές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση και όχι να ανακοινώνονται απλά σε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένους μηχανισμού. και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την στατιστική διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι αμιλητέο. Πάντα γίνονταν συστάσει από τον συμβουλευτικό φορέα, οι οποίε και απορρίπτονταν σε εθνικό επίπεδο, γιατί λέγανε ότι δεν θέλουμε ε, διατάξεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιλάμε για σημαντικές ε, δραστηριότητε που είναι απαραίτητε σε εθνικό επίπεδο. Πώ είναι λοιπόν ε, η συνεργασία με τα κράτη-μέλη γκρινιάζουν που θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί σας ή μήπω λένε τα εθνικά κράτη-μέλη ότι επιτέλους χρειαζόμαστε, ε, ε, λαμβάνουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ, κάποια στοιχεία τα οποία μας χρησιμεύουν σε εθνικό επίπεδο και τι συμβαίνει στα εθνικά δεδομένα. Πρέπει να παρουσιάζονται με κάποια συχνότητα π.χ. κάθε τρίμηνο. Ή μήπως δεν χρειάζονται τέτοια τακτική αναφορά, τακτική παρουσίαση στοιχείων και μπορούμε να κοιτάξουμε τι γίνεται κατά περίπτωση. Ευχαριστώ, Αντολίν. Ευχαριστώ. Όταν εγκρίθηκε το εξαπλό πακέτο, το six pack, ένα από τα στοιχεία που περιλάμβανε ήταν η θέσπιση κάποιων πλαισίων για τους εθνικούς λογαριασμούς στα κράτη-μέλη. Αρχικά στην Ισπανία οι αυτόνομες περιφέρειες έπρεπε να υποβάλουν τριμηνιαίως τις, ε, τις στατιστικές τους πληροφορίες. Τώρα μετά την οδηγία για τα εσωτερικά δημοσιονομικά πλαίσια θα πρέπει αυτό να γίνεται μηνιαία. Το ίδιο και για την κοινωνική ασφάλιση και το καθεξής. Οπότε βρισκόμαστε σε φάση εκτέλεσης και εφαρμογής του εξαπλού πακέτου και φυσικά διανύουμε μια μεταβατική περίοδο και αυτή είναι η ερώτησή μου. Πώς α, α, συνεχίζεται αυτή η διαδικασία στα κράτη-μέλη. Καταφέρουν τα κράτη-μέλη να, να υλοποιήσουν, να έχουν καταφέρει τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τους στόχους. Άλλος κανείς? Όχι. Οπότε κύριε Βίζαρ, έχετε το λόγο να δώσετε τις τελευταίες απαντήσεις και να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Δεν θα πρέπει να υπερμιβούμε το τι μπορεί να κάνει η υπηρεσία μας. Όπως λέει και ε, το όνομά της, είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ασχολούμεθα με θέματα διακυβέρνησης ε, και όχι να δίνουμε απλά βοήθεια. Αλλά πάντως αυτό κάνουμε και είμαστε ακριβώς εξωστρεφείς για να μπορούμε να το κάνουμε. Κάποια από τα θέματα που θέσατε είναι σημαντικά. Αν με κλειδώσετε σε ένα δωμάτιο, μου δώσετε ένα χαρτί και μου πείτε γράψτε εσύ το σωστό πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, θα σας έδινα κάτι το οποίο δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Uh, είναι ένα σύστημα περίπλοκο, με ε, θα έλεγα ε, πολλαπλές αμφίδρομες συνδέσεις ανάμεσα σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Θα είχα ένα υψηλότερο επίπεδο επίσημης ανεξαρτησίας των Εθνικών Στατιστικών Ινστιτούτων ή Αρχών θα είχα το ίδιο επίπεδο αναφοράς ε, στα εθνικά κοινοβούλια, όπως ισχύουν και στα εθνικά κοινοβούλια για τις κεντρικές τράπεζες. Βέβαια μπορεί να συζητάει κανείς τα προβλήματα γενικά ευθύνης ε, σε εθνικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι το σύστημα δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο και αυτό είναι το κομμάτι της διακυβέρνησης. Κάποιοι θα πούν Κύριε Βίζε, μπορείτε να συνεχίσετε να ονειρεύεστε. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε κάποιους στόχους και δεν θα πρέπει να καταφλιβόμεθα εάν δεν τον πετύχουμε το στόχο αυτό το επόμενο έτος. Αλλά πρέπει να έχουμε το όραμα. Παρά το G που περιλαμβάνεται στην εντολή μας και στον τίτλο μας, Νομίζω ότι και η παραγωγή των στατιστικών μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική μέσω της αποφυγής επαναλήψεων, επικαλύψεων, ε, ανταλλαγών, έχοντας κοινούς κανόνες για τον τρόπο παραγωγής των δεδομένων και αναφέρθηκα σε ορισμένους από τους τομείς τους οποίους πιστεύω ότι οι διαφοράς που ισχύουν σε νομικό επίπεδο στα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να οδηγούν σε, διαφορετική, σε διαφορετικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι πιθανές αλλαγές και βελτιώσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης θα συμβαδίσουν και με την βελτίωση των στατιστικών και με τη συγκρισιμότητα των στατιστικών και με την ποιότητα της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων αυτών που είναι υπεύθυνοι. Οι διαφορές τις οποίες αναφερθήκατε δεν είναι μόνο διαφορές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε και προσθέσετε τα ισοζύγια πληρωμών, 190 χωρών στον κόσμο, θα περιμένατε να φτάσουν στο μηδέν. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο πλανήτης ε, αυτή τη στιγμή έχει ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών που είναι 2 ή 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι λίγο θέματα για τα οποία δεν είμαστε βέβαιοι. Πάντως το θέμα της βελτίωσης, της περιοδικότητας, των, της παροχής δεδομένων και της παραγωγής δεδομένων και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν γνωρίζω σε ποια φάση εφαρμογής βρισκόμαστε στα διάφορα κράτη-μέλη οι διαφορές ε, στην πρακτική μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Ανάλογα με το ποιες εσωτερικές ή περιφερειακές ή ομόσπονδες αρχές ανακράτως έχουν τον τρόπο να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς ίσως δεν γνωρίζω ακριβώς το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, αλλά γνωρίζω ας πούμε τις προσπάθειες της Ισπανικής κυβέρνησης, την οποία συνεχάριμεν και η οποία προσπαθεί να βελτιώσει την συλλογή, την επαλήθευση και την διάδοση των εθνικών στατιστικών δεδομένων. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα και μας κάνουν όλους να προβληματιστούμε και με πήραν, εγώ θα επανέλθω σε στατιστικές τροπολογίες για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει ε, σήμερα το απόγευμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε στη δική μας πρόταση να συμπεριλάβουμε και τις περιφερειακές παραμέτρους η ροή των στοιχείων δεν έρχεται τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσαμε γενικότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει από ό,τι φαίνεται υπάρχουν βελτιώσεις και υπό το φως των υποσχέσεων που δόθηκαν στα πλαίσια του εξαπλού πακέτου νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε ότι σημειώσαμε πρόοδο. Αν έχετε περισσότερες ιδέες θα είμαστε πάντα εδώ για να τις ακούσουμε. Ο αριθμός των στατιστικών φακέλων αυξάνεται συνεχώς που έρχονται σε μας και κάποιες ιδέες για τη σωστή τους επεξεργασία είναι χρήσιμες. Θα σας ξαναζητήσουμε να έρθετε εδώ σε ένα χρόνο περίπου ή και νωρίτερα, πέρα της συνεδρίασης.